So, colleagues, we have a very long vote, so please sit down. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολλές ψηφοφορίες, οπότε καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε.